με πληροφορούν περί της εκλογής του κυρίου Δαμιανού Ζοφόλη από 18 Φεβρουαρίου 2015, ο οποίος αντικαθιστά την κυρία Αλεσάνδρα Μορέτη. Το Κοινοβούλιο λαμβάνει υπόψη την εκλογή του νέου συναδέλφου, τον καλωσορίζω και υπενθυμίζω ότι υπόκειται πλέον